Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Παναγία των Παρισιών ήταν ε, ο πρώτος καθεδρικός της ζωής μου. Ως πολίτης των Παρισιών, ως Ιταλός, ως Ευρωπαίος. Αισθάνομαι πληγή βαθιά στην καρδιά μου όπως αισθάνονται όλοι. Ύστερα από τα χθεσινά γεγονότα στο Παρίσι. Στεκόμαστε στο πλευρό των Γάλλων, στο πλευρό της Γαλλίας. Η πληγή αυτή δεν πρόκειται να σβήσει γρήγορα. Πρέπει όλοι μας να στρατευτούμε και δεχόμενο την πρόταση ενός συναδέλφου ευρωβουλευτή που μου πρότεινε να κάνουμε ε, έρανο όλοι για να στηρίξουμε την Παναγία των Παρισίων θα φροντίσω να τοποθετηθεί ένα κοιτίο εράνου έξω από την αίθουσα ώστε να καταθέσουμε και προτείνω να καταθέσουμε τη σημερινή μας αποζημίωση όλοι ε, για να ξαναχτιστεί ό,τι μπορεί να ξαναχτιστεί από, αυτή την, ε, από αυτό το κτίριο, από ε, τον Καθεδρικό Ναό, ως μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πυροσβέστες, τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Γαλλίας, που χτες έκαναν μάχη σκληρή, έδωσαν μάχη σκληρή κατά της φωτιάς που κατέστρεφε το καθεδρικό ναό. Στηρίζομαι στη βοήθειά σας και ελπίζω το μήνυμα αυτό από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζω και από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου να είναι ένα μήνυμα το οποίο θα πουλώσει τι πληγέ τη Γαλλία, των Γάλλων, όλου του Ευρωπαϊκού, όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Σα ευχαριστώ. La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca dichiarazione del Ξεκινάει η μερίσια διάταξη. Έχουμε κοινή δήλωση Συμβουλίου και Επιτροπής ε, για την έκβαση του Συνόδου Κορυφής της ε, προηγούμενης εβδομάδας, 10 Απριλίου, για την ε, αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ξεκινήσει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Ντόναλτ Τούσκ, στον οποίο και δίνω το λόγο. Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, από τη θέση αυτή θα ήθελα να εκφράσω την ε, συμπαράστασή μου και την ελεγγύη μας ε, προς το γαλλικό λαό για την τραγωδία που αντιμετωπίζει και αυτό όχι ως ε, πρόεδρος μόνο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και ως πολίτης του Κτάνσκ που κατά 90% είχε καεί και καταστραφεί στον πόλεμο θα ξαναχτίσετε την Παναγία των Παρισίων, θα την ξαναδείτε και καλό και τα 28 κράτη-μέλη να συμβάλλουν προς το στόχο της ανοικοδόμησης. Είμαι βέβαιος ότι η Γαλλία μπορεί να το καταφέρει μόνο, μόνη της αυτό. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ περισσότερο από την παροχή υλικής βοήθειας. Η πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων μας ε, κατέστησε απόλυτα σαφές ότι μας ενώνει κάτι πολύ πιο σοβαρό και πιο βαθύ από κείμενα συνθήκων. Έχουμε κάτι κοινό και το αναγνωρίζουμε αυτό όταν βλέπουμε τι μπορούμε να χάσουμε και όταν αντιλαμβανόμαστε ότι θέλουμε να το υπερασπιστούμε όλοι μαζί. Την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 27 Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων σε συμφωνία και με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου χορήγησε μια παράταση ευέλικτη της περίοδου που προβλέπει το άρθρο 50 έως την 31η Οκτωβρίου του 2019. Πρόκειται για μια παράταση η οποία επιτρέπει περισσότερο χρόνο, χορηγεί περισσότερο χρόνο και ευελιξία στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για να βρει μια δέξοδο από την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και ελπίζω να την αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει ένα σαφές μήνυμα από το Ηνωμένο Βασίλειο για τα περαιτέρω. Και αν κυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης, η περίοδος παράτασης αυτομάτως λύγει την πρώτη ημέρα του μήνα που θα ακολουθεί την ανακοίνωση της κύρωσης και άρα από εκείνη τη μέρα θα έχει αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να είναι απολύτω σαφέ ότι δεν πρόκειται να ξανανοίξει η συζήτηση για τη Συμφωνία Αποχώρησης. Ωστόσο, προκειμένου να διευκολυθεί η διαδικασία απόχώρηση οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διατεθειμένοι να ξανασυστήσουν την πολιτική διακήρυξη για τη μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον προχωρήσουν οι θέσεις ε, του Ηνωμένου Βασίλειου. Την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άλλαξε ε, λογική σε σχέση με τη χορήγηση μιας πιο ήπιας παράτασης ε, για το Ηνωμένο Βασίλειο στην χορήγηση μιας μακρύτερης παράτασης, χρονικά μακρύτερης δηλαδή, πράγμα το οποίο και εγώ προτιμούσα για να είναι πιο επικοδομητική. Αυτό επιτρέπει την διατήρηση κάθε επιλογής, δηλαδή και την κυρίωση της υφισταμένης συμφωνίας αποχώρησης και την, τον αναλογισμό των συνθήκων και της επιλογής του Brexit, εφόσον το επιθυμεί ο Βρετανικός λαός. Επίσης, ε, με την παράταση αυτή μπορεί να δοθεί έμφαση και σε άλλες προτεραιότητες εξίσου σημαντικές που έχουν να κάνουν και με τις εμπορικές συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, με, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συγγνώμη. Επίσης, ε, ξέρω ότι ορισμένοι μπορεί να έχουν διατυπώσει ανησυχίες πως το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να έχει παρελκυστική και παρεμποδιστική τακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, από εδώ και εμπρό με την παράταση αυτή. Ωστόσο δεν θελήσαμε να ακούσουμε αυτές τις φωνές και τις κασάνδρες και ε, θεωρούμε ότι η στάση μέχρι τώρα του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν και θα συνεχίσει να είναι η στάση ενός υπεύθυνου ε, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε κανένα λόγο να θεωρούμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Επίσης αυτή η παράταση και αυτή είναι η τρίτη θέση μας, ε, επιτρέπει να μην υπάρξει καθυστέρηση στην ε, διαδικασία της ολοκλήρωσης του Brexit που θα κρατήσει περισσότερο από έξι μήνες. Δηλαδή θα έχουμε περισσότερη βεβαιότητα για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες για την εξέλιξη του Brexit. Μία από τις συνέπειες αυτής της συμφωνίας είναι ότι τον επόμενο μήνα στον Ηνωμένο Βασίλειο θα δεξαχθούν ευρωεκλογέ. Πρέπει αυτή την προοπτική να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα. Τα μέλη, οι Βρετανοί βουλευτές του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις για, το, για αρκετούς μήνες τουλάχιστον μετά τις ευρωεκλογές και αυτό ήθελα να το αναφέρω σήμερα διότι ε, αντετάχθην στην ιδέα που κυκλοφορούσε σε περίπτωση παράτασης το Ηνωμένο Βασίλειο να τύχει μεταχείρισης δεύτερης κατηγορίας μέλους. Αυτό το απορρίπτω λοιπόν και σας παρακαλώ και εσάς, εάν τυχόν και ακουστούν τέτοιε ιδέες εδώ στο Κοινοβούλιο, να τις απορρίψετε ανεπιφύλακτα. Και γνωρίζω ότι και από τις δύο πλευρές της μάχης, από τις δύο όχθες της μάχης, όλοι μας εγώ προσωπικώς, είμαστε εξαντλημένοι από αυτή την ιστορία και το καταλαβαίνουμε, είναι απολύτως κατανοητό. Πλην όμω αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για να πει κανεί. άντε ας το κλείνουμε το θέμα, γιατί κουραστήκαμε μόνο και μόνο. Όχι, πρέπει να συνεχίσουμε το Brexit να το αντιμετωπίζουμε με πνεύμα ανοιχτό και τρόπο πολιτισμένο, διότι ό,τι και να συμβεί, το πεπρωμένο μας είναι κοινό θα είμαστε πάντα συνδεδεμένοι και θέλουμε να παραμείνουμε στενοί φίλοι και εταίροι και στο μέλλον. Κατά την ε, σύνοδο κορυφής ένας από τους ηγέτες μας είπε ότι δεν πρέπει να ονειροπολούμε και δεν πρέπει να θεωρούμε ότι μπορεί να αναστραφεί το Brexit. Απάντηση δεν έδωσα εκείνη τη στιγμή. Σήμερα όμως και ενώπιον ημών θέλω να πω πως σε αυτή τη δύσκολη στιγμή στην ιστορία μας Χρειαζόμαστε ονειροπόλους, χρειαζόμαστε όνειρα. Δεν μπορούμε να υποκύψουμε στην μυρολατρεία. Τουλάχιστον για μας που θέλουμε μια καλύτερη και πιο ενωμένη Ευρώπη. Αγαπητοί φίλοι, πρόκειται για τελευταία συνεδρίαση που θα συναντηθούμε σε αυτή σας την βουλευτική περίοδο. Ελπίζω να έχω τη χαρά να σας ξαναδώ, τους περισσότερους από εσάς τουλάχιστον, μετά τις εκλογές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ζωάν Juncker. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χθες ήταν μια πολύ δυσάρεστη μέρα για όσους αγαπούν τη Γαλλία και το Παρίσι. Στη ζωή όλων μας, το Παρίσι δεν είναι ένα τυχαίο μέρος είναι μια πόλη όπου όλοι θέλουμε να πάμε για να ξαναρωτευτούμε. Και το να διαπιστώνουμε ότι το Παρίσι υφίσταται μια τραγωδία που δεν είναι μόνο αρχιτεκτονική, αλλά αφορά τη ζωή όλων των Γάλλων. Να βλέπουμε οι φωτιές να καταστρέφουν το εξωτερικό σύμβολο της δύναμης της Γαλλίας γιατί πάρα πολλοί επισκέπτονται την ε, Παναγία των Παρισιών, την Notre Dame Όλα αυτά μας λείπουν ιδιαίτερα. Ε, ένα σημαντικό σύμβολο της Γαλλίας υπέστη μια σοβαρή πληγή και είμαστε όλοι μόνοι. Έχουμε όλοι πληγή από αυτό το γεγονός και εκφράζω την πλήρη συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ήδη διακήρυξε ότι θα βοηθήσει όλες τις προσπάθειες που κάνει ε, η Γαλλία, ε, το Παρίσι, η Γαλλία, η Ευρώπη, όλοι επλήγημεν και εκδηλώνουμε την αλληλεγγύη μας με τους Γάλλους φίλους. Since uh, Από τότε που ολοκληρώθηκαν εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ ίδιος περιμένουμε να ολοκληρωθεί το Brexit. Βεβαίω πρέπει να εστιάσουμε και σε πολλά άλλα θέματα. Στο θετικό θεματολόγιο που έχουμε εντοπιό μα. Και γι' αυτό θέλω να είμαι πολύ σύντομο. Την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο έλαβε μία ε, ενιαία, ενωμένη και υπεύθυνη απόφαση για να παραταθεί η περίοδο εφαρμογή του άρθρου 50 μέχρι 31 Οκτωβρίου τρέχοντο. Αυτή ήταν μία αποδεκτή λύση για τρει λόγου. Πρώτα απ' όλα, και με τη στήριξη του σώματός σας εγκρίναμε όλα τα αναγκαία έκτακτα μέτρα και είμαστε έτοιμοι να υπάρξει, εάν υπάρξει συμφων... Ε, ε, Brexit χωρίς συμφωνία, αλλά η Ένωσή μας δεν έχει να κερδίσει τίποτα από την ε, σοβαρή ανταραχή που θα προκληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτοί που θα επωφεληθούν είναι αυτοί που είναι κατά της διεθνούς συνεργασίας και θέλουν να υπονομεύσουν τη διεθνή τάξη. Και ποτέ ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να διώξουμε ένα μέλος μας. Δεύτερον, προστατεύσαμε την ακυρεότητα και τη λειτουργία και του σώματό σα και όλων των θεσμικών οργάνων. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να είναι μέλο τη 23 Μαου, τότε πρέπει να διεξαχθούν και εκεί ευρωεκλογέ. Αν δεν το κάνει και αν δεν έχει επικυρωθεί η συμφωνία αποχώρηση μέχρι τι 22 Μαου, η παράταση θα λήξει στις 31 Μαΐου. Αυτή είναι η κατάσταση από πλευράς ε, νομικής κατάστασης. Επίσης, διασφαλίσαμε ότι δεν χρειάζεται να συζητούμε το Brexit ε, κάθε 15 ημερών. Και δώσαμε στον Ηνωμένο Βασίλειο το χρόνο και το περιθώριο για να ξεπεράσει το αδιέξοδο. Όταν θα αρχίσει να ισχύει η Συμφωνία Αποχώρησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί όσο γίνεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως κατά τη διάρκεια ε, των διαπραγματεύσεων για τον Brexit. Η πλήρης διαφάνεια των διαπραγματεύσεών μας και η στενή και αποτελεσματική συνεργασία με την ομάδα Brexit του Κοινοβουλίου ήταν η ισχύ μα κατά τι διαπραγματεύσει και θέλουμε αυτέ οι καλέ πρακτικέ να συνεχιστούν και κατά την εφαρμογή τη συμφωνία αποχώρηση. Οποτεδήποτε θα πρέπει να ληφθούν αποφάσει σε αυτή την λεγόμενη κοινή επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φροντίσει να συμμετέχει πλήρω στο Κοινοβούλιο και θα λάβει ιδιαίτερα υπόψη τι απόψει του. Μάθαμε να προσέχουμε ιδιαίτερα αυτά που συμβαίνουν στην Βουλή των Κοινοτήτων τους τελευταίους μήνες. Αλλά θέλω να είμαι απόλυτα σαφής για τον Brexit. Τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί εναντίον των αποφάσεων αυτού του οίκου της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για τον Brexit χωρίς να ληφθούν πλήρως υπόψη οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι, στις 31 Οκτωβρίου θα λήξει η νέα προθεσμία για μία συντεταγμένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και αν δεν έχει επικυρωθεί από το Βρετανικό Κοινοβούλιο μέχρι τότε η συμφωνία αποχώρηση, θα υπάρξει ένα σκληρό Brexit που όλοι θέλουμε να αποφύγουμε. Φυσικά, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αποφασίσει επίση να αποσύρει την αίτηση αποχώρηση. Αυτό το είπε σαφώ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά αυτή δεν είναι η υπόθεση εργασία μου. Όπω επίση δεν είναι ότι θα υπάρξει καμία παράταση μετά την 31η Οκτωβρίου. Δεν είναι η υπόθεση εργασίας μου, ούτε αυτή. Δεν μου αρέσει αυτή η ημερομηνία 31 Οκτωβρίου. Κατά τα άλλα δεν μου αρέσει λοιπόν. Γιατί είναι η τελευταία μέρα της θητείας μου ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και δεν μπορεί να γίνει λοιπόν για αυτό το λόγο καμία νυχτερινή ε, συνεδρίαση. Γιατί στις 12 η ώρα θα πρέπει να αποχωρήσω εγώ. Αλλά μπορεί να παραμείνει ο Ντόναλτ Τούσκ. Ε, έγινα πρόεδρος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί ήθελα να επιταχύνω τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θεωρούσα ότι έπρεπε να γίνουν περισσότερα για την κοινωνική Ευρώπη. Κάναμε περισσότερα, αλλά όχι επαρκή. Επίσης, Ήθελα να γίνουν οι αναγκαίε μεταρρυθμίσει τη ε, Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Θα ήθελα για τη χρηματοδότηση τη επόμενη περίοδου 21-28 να είχαμε συμφωνήσει. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι πολλοί νέοι, οι πολλοί ερευνητέ, οι φοιτητέ που απολαμβάνουν ε, ε, ενισχύσει από το έρασμος να ε, υποστούν τις συνέπειες του Brexit. Δεν τους αξίζει κάτι τέτοιο. Πρέπει να φροντίσουμε ούτω ώστε να μην απομακρυνθούν από την Ευρώπη. Τώρα προς τα πού θα πάει το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό θα το αποφασίσει το Λονδίνο. Και όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα. Χαιρετίζω ιδιαίτερα το ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση τώρα βρίσκονται σε ε, διαπραγματεύσεις. Αυτό το χαιρετίζουμε ως πρόοδο. Και ε, στο βρετανικό πλαίσιο βέβαια είναι πρόοδος, αλλά δεν είναι φυσιολογικό. Το ότι οι κύριες δυνάμεις τόσο αργά αποφασίζουν να συνοηθούν, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Και χαιρετίζω το ότι επιτέλους τώρα γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις. Το πότε θα αποχωρήσουν από το Ηνωμένο Βασίλειο Βρετανή είναι δικό του θέμα. Το πότε και το πώς. Και βεβαίως ε, συμφωνήσαμε για μια συμφωνία αποχώρησης ε, τον Νοέμβριο του 2018. Αυτό το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του περασμένου Νοεμβρίου εξακολουθεί να ισχύει. Σε καμία ε, περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε επιπλέον διαπραγματεύσεις πάνω στη συμφωνία αποχώρησης. Για την πολιτική διακήρυξη για το μέλλον ε, των σχέσεων, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, αν εκφραστεί επιθυμία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, το Brexit δεν είναι το μέλλον της Ένωσης. Το μέλλον της Ένωσής μας είναι πολύ περισσότερο από το Brexit. Το Brexit δεν πρέπει να δυσχεράνει τις εργασίες μας για τις μεγάλες προτεραιότητές μας. Γι' αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε επί δύο αρχών. Πρώτον, όσο είναι μέλος του Ηνωμένου Βασίλειου υπολογίζουμε ότι θα είναι υπεύθυνη, έντιμη η συνεργασία μαζί του. Είναι αρχή. Είναι βασική αρχή της συνθήκης που πρέπει να γίνει σεβαστή. Δεν ε, υπολογίζουμε, απαιτούμε να υπάρξει υπεύθυνη και έντιμη συνεργασία. Δεύτερον, δεν υπάρχει κράτο μέλο δεύτερη κατηγορία. Αλλά ένα κράτο μέλο θέλει να αποχωρήσει από την Ένωση, 27 άλλοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συνεδριάζουν χωριστά για τα θέματα του μέλλοντο τη Ένωση. Δεν είναι αυτό καινοτομία. Το Δεκέμβρη του 1997 ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ω πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ξεκίνησε το Eurogroup κατά της άποψης των Βρετανών, των Σουηδών, των Δανών και κάποιων άλλων. Το Eurogroup είναι μια περιορισμένη μορφή συνεδρίασης για όσους ενδιαφέρονται για την οικονομική οικοδόμηση της Ένωσης και την νομισματική. Είχαν το δικαίωμα να συνεδριάζουν και συνεδριάζουν και τα αποτελέσματα είναι ουσιώδη. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει στρατηγικές προκλήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί. Πρώτα απ' όλα, στο Σύμπιου το Μάιο θα συζητήσουμε τις στρατηγικές μας κατευθύνσεις για τα επόμενα χρόνια. Και κατόπιν έχουμε και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, επί του οποίου, επί της αρχής, πρέπει να αποφασιστεί τον Οκτώβριο και πρέπει να εκλεγεί η επόμενη ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου το εκλογικό σώμα είναι το μεγαλύτερο μετά από αυτό τη Ινδία. Και πρέπει να εκλέξουμε και μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει τον επόμενο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το μέλλον τη ενωσή μα έχει να κάνει και με τη θέση μα στον κόσμο. Γιατί έχουμε εμπορικέ συμφωνίε. Πρέπει να δούμε τη σχέση μα με του μεγάλου διεθνεί εταίρου μα, ιδιαίτερα με την Κίνα, με την οποία την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση κορυφή και τον ε, προσεχή Ιούνιο στην Όζακα θα συνεδριάσει το G20, όπου θα συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον του παγκοσμίου εμπορίου. Όλα αυτά είναι πραγματικά πιο ουσιώδη από τα επεισόδια που σχετίζονται με τον Brexit. Η Ευρώπη συνεχίζει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να θυμίσω στους συναδέλφους ότι στη διάρκεια αυτού του Συμβουλίου εγώ επέμεινα για την αξιοπρέπεια του Κοινοβουλίου, για το ρόλο που έχει. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως ταξί και οι διαπραγματεύσει για το Brexit θα πρέπει να λάβουν υπόψη το ρόλο του δικού μας θεσμού. Νομίζω πως αυτό είναι για μας προτεραιότητα και πιστεύω πως μιλώ εξ ονόματος όλων των συναδέλφων γιατί είμαστε το πρώτος θεσμός στη συνθήκη και ε, θεωρούμε ότι πρέπει όλα τα 28 κρατη να σέβονται το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, ο κύριο Γκονζάλη Πόνς έχει τώρα το λόγο. Θα πρέπει να πω τον πόνο που ένιωσα εχθέ όταν έβλεπα να καίγεται η καθεδρική τη Νότρε Η πυρκαγιά αυτή μα έχει επηρεάσει όλους αν ήμασταν Γάλλοι. Όλοι αισθανόμαστε θλίψη το ίδιο αποσβολωμένοι ε, και αδύναμοι και σήμερα το πρωί όλοι θέλουμε να ξεκινήσουμε την ανοικοδόμηση. Οι λαοί δεν αναπτύσσονται όμως κλαίγοντας μαζί, αλλά προχωρώντας μαζί. Και η χθεσινή πυρκαγιά της Νοτριντά μας κάνει περισσότερο Ευρωπαίους, όχι επειδή κλάψαμε μαζί, αλλά επειδή μαζί θα ανοικοδομήσουμε την, ε, τον καθεδρικό ναό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει οικονομική βοήθεια και τεχνίτες, όλους ε, όσοι είναι απαραίτητοι για να ξαναχτιστεί ο καθεδρικός ναός όπως χτίζονταν και στο παρελθόν ακριβώς οι καθεδρικοί ναοί, καλώντας όλους να συνεργαστούν για ένα τέτοιο όραμα. Η χθεσινή πυρκαγιά έδειξε πως οι Ευρωπαίοι δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας. Η Ευρώπη είναι η απάντηση στη φωτιά, στην καταστροφή, στον εγωισμό και στην φτώχεια. Γι' αυτό ε, χτες το βράδυ βλέποντας να καίγεται ο καθεδρικός ναός αναρωτήθηκα ακόμα μια φορά ε, μα γιατί θέλουν να φύγουν από εδώ οι Βρετανοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα αξιών και αρχών. Εάν το, μας φαίνεται πως δεν λειτουργεί ε, θα πρέπει να τη μεταρρυθμίσουμε για να λειτουργήσει καλύτερα. Αλλά δεν φεύγεις, δεν φεύγεις γιατί οι αξίες είναι κοινέ, παραμένουν κοινέ και σε καμιά περίπτωση δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Ό,τι και αν γίνει Τρία διδάγματα πρέπει να αποκομίσω από το Brexit. Πρώτον, ότι στην πολιτική δεν μπορεί κανεί να υποσύσχεται αυτό που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει. Δεύτερον, στην πολιτική τα ψεύδη πάντοτε φέρνουν ε, απογοητεύσει. Και έπειτα οι δεσμοί που χτίζει η ιστορία δεν μπορούν να καταλύονται μόνο και μόνο από, λόγω εγωισμού. Το Brexit είναι κάτι το αόριστο και χωρίς ημερομηνία. Για μένα η Ευρώπη είναι ολοκληρωμένη. Ε, δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν οι πολιτικοί οι Βρετανοί όμως δεν μπορούν να βρουν λύση, ας δώσουν το λόγο πάλι στο λαό. Έπειτα η πυρκαγιά της Νοτραντάμ μας δείχνει και πάλι ότι μιλάμε υπερβολικά πολύ για το Brexit και πολύ λίγο για όλα τα υπόλοιπα. Λυπάμαι για την ματαιοδοξία των Βρετανών πολιτικών. Όμως σήμερα η θλίψη για την πυρκαγιά της Νότρεντάμ με καθιστά ακόμα περισσότερο Ευρωπαίο παρά η απογοήτευσή μου λόγω της ανικανότητας. Ευχαριστώ εκ μέρους της, της Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ο κύριος Ούντο Μπούλμαν έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα το πρωί ενωμένοι κοιτάμε και στρέφουμε το βλέμμα προς το Παρίσι. Και θέλουμε να πούμε είμαστε η Νότρο Θέλουμε να πούμε Παρίσι δεν είσαι μόνος σου. Γαλλικέ λαέ δεν είσαι μόνος σου. Έτσι εκδηλώνουμε εμείς την ε, Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Και με αυτό το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης οφείλω να συγχαρώ εσάς, Πρόεδρε Τάσκ, τους που αναλάβατε εσείς την ευθύνη να χορηγήσετε την παράταση στο Ηνωμένο Βασίλειο για το Brexit, γιατί έτσι αποφύγατε την κατάρρευση, την σύγκρουση. Ποιος θα την πλήρωνε την κατάρρευση αυτή, τον κατακριμνισμό αυτών, ούτε η πολιτικοί, ούτε κανείς άλλος από τους μεγάλους και ισχυρούς, αλλά οι πολίτες αυτοί οι οποίοι μπορεί, μπορούν να ελπίζουν μόνο στο να βρούνε μια καλή δουλειά στο ένα ή το άλλο κράτος, αυτό που τους επιτρέπει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ανοιχτά σύνορα. Και παίξατε με τη μοίρα των πολιτών της χώρας. Ας το απέφυγαν λοιπόν χάρη στον πρόεδρο Γιουνκέρ, χάρη στον πρόεδρο Τούσκ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τους υπεύθυνου πολιτικούς που έλαβαν την απόφαση της παράτασης. Και θα ήθελα να σας ε, επικροτήσω επίσης πρόεδρε Τούσκ όταν ε, είπατε ότι έχει δικαιώματα όπως κάθε κράτος μέλος όσο παραμένει μέλος και αυτό ισχύει και για του βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν μιλούμε για μικροκομματικά ζητήματα ή επιλογές. Μιλούμε για αξιοπρέπεια του κάθε ψηφοφόρου της εκλογικής περιφέρειας, του κάθε εκπροσωπουμένου εδώ και βεβαίως θα καλωσορίσουμε τους εκλεγμένους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Ηνωμένο Βασίλειο και θα έχουν κάθε ε, δικαίωμα και υποχρέωση και στη δική μου την πολιτική ομάδα εντασσόμενη σε κάθε περίπτωση. Και είμαι πεπισμένος ότι και μετά την 31η Οκτωβρίου θα ανοίξει μια νέα συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα αποτελέσει το έναυσμα του τέλους του Brexit. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Γιατί εν τέλει θα έχουν την ευκαιρία οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου να μιλήσουν, να εκφράσουν τη γνώμη τους το Κοινοβούλιο, το Βρετανικό, δεν μπορεί να λάβει απόφαση. Σε τέτοιε περιπτώσει είμαι πεπισμένο ότι πάντα, πάντα πρέπει κανεί να στρέφεται στην ετοιμιγορία του λαού. Και ό,τι είναι στραβό να βγει από τη συζήτηση. Να παραμείνει ό,τι είναι σωστό. Το take back control σημαίνει δίνουμε το λόγο στο λαό, όχι στο δρυμερή διάλογο. Και είμαι πεπισμένο για το ότι το Brexit δεν αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Brexit δεν αφορά καν μόνο όλους αυτούς που θέλουν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit σημαίνει πολύ περισσότερα πράγματα. Έχει να κάνει με τους Πούτιν, με τους Τραμπ, με τους Στιβ Μπάνον, με τους Σαλβίνι που προσπαθούν να καταστρέψουν αυτά που έχτισαν ο Ρομπέρ Σουμάν και ο Ζαμονέ. Αυτά τα οποία ο Νάουερ και ο Βίλι Μπραντ οραματίστηκαν όλα αυτά τα οποία είναι κοινά και αυτά για τα οποία ακριβώς και θα υπερασπιστούμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αποτελεί τη σωστή απάντηση στα μεγάλα ερωτηματικά για το μέλλον. Και βλέπουμε ποια είναι η απάντηση και στη Φινλανδία την είδαμε και στη Σουηδία τη βλέπουμε. Οι άνθρωποι θέλουν να αντιμετωπίσουν τους ακραίους δεξιούς και ενώνουν τις δυνάμεις τους και ελπίζω να δώσει την αντίστοιχη απάντηση με αυτή που δίνουμε εμείς και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εκεί όπου στην Ανδαλουσία ή όπου αλλού έχει περιφερειακή περιφερειακές, τοπικές, ευρωπαϊκές, εθνικές εκλογές και στην Ιταλία και αλλού ανάλογα με το με ποιον θα συμμαχίσει θα κρυθεί η απάντηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι τασόμαστε στην Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές της Ευρώπης, ο κύριος Καμάλ. Κύριε Πρόεδρε, όταν βλέπει κανείς τις εικόνες ε, χθε που και εγώ ήταν η Νότρονταμ, είναι, ε, σκέφτεται ότι πρέπει να αφήσουμε την πολιτική κατά μέρο όπου και αν είναι, από όπου και αν είναι κανεί Βρετανό, από την Ευρώπη, από τον υπόλοιπο κόσμο, όλοι εθλίψαν βαθιά. Πριν από 25 χρόνια η γυναίκα μου σπούδαζε στη Γαλλία και για ένα διάστημα εργαζόταν στη, στο Παρίσι και επισκεφθήκαμε την Ντάμ που είναι ένα σύμβολο και την προηγούμενη εβδομάδα ξαναπήγαμε. Πήραμε φωτογραφίε. Σκεφτείτε τα εκατομμύρια που επισκέφθηκαν ε, αυτή την εκκλησία ανεξάρτητα από την πίστη τους είναι σύμβολο όχι μόνο του Παρισιού αλλά της ιστορίας της Ευρώπης αλλά ολόκληρου του κόσμου και ναι εγώ ε, δεν είμαι αυτή τη πίστεως αλλά συμμερίζομαι τον πόνο σας εδώ σε αυτήν την αίθουσα και ελπίζω όλοι να συνεργαστούμε είτε Βρετανοί είτε Ευρωπαίοι είτε από πέρα από την Ευρώπη για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πανικοδομηθεί. Πολλοί ελπίζαμε ότι δεν θα γινόταν αυτή η συζήτηση σήμερα και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει αποχωρήσει στι 29 Μαρτίου ή ακόμη και την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε με την κατάσταση όπω έχει. Η Βρετανική κυβέρνηση είναι ακόμη δεσμευμένη να υπάρξει συντεταγμένο Brexit και αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ω να τον πιο σύντομα. Αυτό ο στόχο τη, ούτω ώστε οι λαοί και των δύο πλευρών να εστιάσουν στο μέλλον. Αυτό που ανέφερε ο Ζαν Κλοντ Το θετικό θεματολόγιο. Ωστόσο, καταλαβαίνω ότι η υπομονή σα ε, έχει φτάσει στα ωριά τη. Και πραγματικά αναρωτιέστε τι συμβαίνει στο Westminster. Αλλά η συμμετοχή στην Ένωση έχει προκαλέσει ε, διχόνοια στη χώρα μου σε πολλά, για πολλά χρόνια. Όχι μόνο στο δικό μου κόμμα, αλλά και στο κύριο κόμμα τη αντιπολίτευση. Και αυτέ οι διχόνοιε βλέπετε ε, πώ εξελίσσονται και τι ρόλο παίζουν. Και πολλοί ρωτάνε γιατί δεν συζητήσατε τι διακομματικέ συναντήσει νωρίτερα. Και μπορεί να φαίνεται φυσιολογικό για ορισμένου από τι χώρε τη δικέ σα, αλλά δεν λειτουργεί έτσι το κοινοβουλευτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Κοιτάξτε τη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου τα δύο κόμματα ε, κάθονται το ένα απέναντι από το άλλο. Όχι στο πλάι, όπω εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο. Από τη μία πλευρά είναι η κυβέρνηση, από την άλλη η αντιπολίτευση. Και αντί να προσπαθούν να φτιάξουν ε, συνεργασίε, είναι πολύ πιο αντιπαραθετικό το σύστημα. Οι συζητήσει αυτέ που γίνονται τώρα δημιουργούν, ε, δημιουργούν συναισθήματα άβολη κατάσταση και από τι δύο πλευρέ. και σε μένα τον ίδιο. Η απάντηση λοιπόν που δόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα τη παράτασης δεν είναι ίσως η ε, απάντηση που ήθελαν όλοι, αλλά είναι μια προσπάθεια να επιδιωχθούν άλλε λύσει. και ελπίζω οι συνάδελφοί μου στο Westminster να μην χρειαστεί να πάρουν πολύ χρόνο. Η οικονομία μα, η πολιτική μα ζωή και η χώρα μα χρειάζονται βεβαιότητα. Στόχο μα πρέπει να είναι να βρούμε μια λύση που θα μα επιτρέψει να αποφύγουμε τη συμμετοχή σε ευρωεκλογέ. Ήρθε τώρα η ώρα για πραγματι... πραγματισμό, για ρεαλισμό. Α το καταφέρουμε. Και κύριε Τούσκ, σα ευχαριστώ για την πιο επικοδομητική σα στάση την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με κάποιε άλλε δηλώσει που είχατε κάνει στο πρόσφατο παρελθόν. Νομίζω ότι τα λόγια σα πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου είχαν το σωστό τόνο. Ότι το θέμα δεν είναι να ε, ταπεινωθεί κανεί ή να υπάρξουν αλληλοκατηγορίε. Πρέπει να παραμείνουμε φίλοι για να προχωρήσουμε στο μέλλον με μια ε, μελλοντική εταιρική σχέση που να διαρκεί. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ε, και σε προηγούμενες καταστάσεις σε δύσκολη θέση, αλλά ε, τα καταφέρνουμε πάντα και ελπίζω ότι και αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε. Και διαρωτώ με αγαπητοί συνάδελφοι, για να πω κάτι προσωπικό. Ίσως είναι η τελευταία μου ομιλία από αυτή την έδρα, σε αυτό το εμικύκλιο μετά από σχεδόν 14 χρόνια. Θέλω να πω ότι ε, είτε συμφωνούσαμε, είτε διαφωνούσαμε, είτε πανεκλεγείτε, ή θα αντιμετωπίσετε νέε προκλήσει. Σα ευχαριστώ όλου ε, για την ε, εργασία σα που συμμετείχατε σε αυτή την καταπληκτική εμπειρία και εύχομαι σε όλου σα καλή τύχη, ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Καμά. Ο επόμενο, ο πρόεδρο τη ε, ομάδα των φιλελευθέρων, Κύριο Γκίφερ Χόστατ. Κύριε Πρόεδρε, όπως και οι συνάδελφοι, και ο πρόεδρος Τούσκ και ο πρόεδρος Γιούνκερ να εκφράσω και εγώ τον πόνο μου για την τρομερή πυρκαγιά χθες βράδυ στο Παρίσι. Είμαι πεπισμένο ότι από κοινού θα ξαναχτίσουμε την Νότο Ντάμ του Παρισίων και θα είναι ακόμη πιο όμορφη με περισσότερη ακτινοβολία από ό,τι στο παρελθόν. Η Παναγία των Παρισίων της Γαλλίας είναι η Παναγία της Ευρώπης. Είμαι πεπισμένος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τούσκ. Ξέρω ότι το κοινοβούλιο μας δεν ε, συμμετείχε στην απόφαση που πήρατε την προηγούμενη Τετάρτη. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας προειδοποιήσω για το εξή. Για τις επιπτώσεις ε, της απόφασης που λάβατε την, την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί μέχρι τώρα υπήρξε ενότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενότητα των 27. Αλλά ενότητα και μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Αυτή η ενότητα βασιζόταν στην εργασία του διαπραγματευτή μας. Θέλω να το υπενθυμίσω αυτό. Ο Μισελ Μπανιέ, τον οποίον θέλω να συγχαρώ για τη θαυμάσια εργασία του. Και αυτή η ενότητα, κατά τη γνώμη μου, κύριε Τάσκ, πρέπει να σας πω ειλικρινά, ότι διακυβεύεται τώρα. Αντί να στείλουμε την κυρία με στο Λονδίνο χωρίς καμία παράταση ή το πολύ με μια πολύ σύντομη, λίγες μέρες, μια εβδομάδα, της δώσατε ένα εξάμεινο. Ένα εξάμεινο. Ξέρετε πολύ καλά ότι στις 31 Οκτωβρίου δεν υπάρχει επαρκή χρόνο για να υπάρξει ουσιώδη αναθεώρηση του Brexit και επίση αρκετά μακριά η 31 Οκτωβρίου για να υπάρχει επίγουσα ανάγκη για δράση. Αυτές είναι οι επιπτώσεις. Βέβαια δεν ε, αποκαλώ την απόφαση αυτή βλακίες, όπως λέει ο κύριος Κόμπερν, ο οποίος ό,τι κάνουμε εδώ πέρα τα λέει βλακίες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Φοβάμαι ότι θα συνεχιστεί η αβεβαιότητα και θα παραταθεί η αναποφασιστικότητα και φοβάμαι ότι θα εισαγάγει τα χάλια του Brexit σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δηλητηριάσει τις επικείμενες ευρωεκλογέ. Περαιτέρω, φοβάμαι ότι... Ξέρετε, υπάρχει μια έκφραση στα Ολλανδικά. Θα κάνει το κοινοβούλιο μας, φοβάμαι, θα το κάνει σαν περιστερεώνα. Δηλαδή οι Βρετανοί θα πετάνε στον περιστερεώνα, μετά θα πετάνε από τον περιστερεώνα και εμείς θα περιμένουμε. πότε θα ε, μπορέσουν αυτοί που επιλέξαμε για να τους αντικαταστήσουν ε, αυτούς που αποχωρούν. Ο Μπάνξι, όπως ξέρετε, έκανε ένα ωραίο σχέδιο που φτιά, ε, εικονίζει το Westminster σαν να είναι γεμάτο με μαϊμούδες και ίσως να κάνει και άλλο ένα που θα κάνει το δικό μας σώμα γεμάτο με περιστέρια. Μια άλλη εικόνα. Φοβάμαι λοιπόν ότι με αυτή την απόφαση η πίεση για να υπάρξει διακομματική συμφωνία, όπως ανέφερε ο κύριος Καμάλ, θα εξαφανιστεί. Και τα δύο κόμματα μπορεί για άλλη μια φορά να επανέλθουν σε αυτό που κάνουν εδώ και μήνες. Να περιμένουν να λήξει προθεσμία. Και η απόδειξη είναι ότι η πρώτη απόφαση που πήρε η πρώτη απόφαση που πήρε μετά από αυτή την τελευταία εξέλιξη το Βρετανικό Κοινοβούλιο ήταν να διακόψει για τις διακοπές του. Δεν περίμενα να ε, το πω αυτό, αλλά ίσως το μόνο που μπορεί να μας σώσει είναι ο Νάιτζολ Φαράτζ. Γιατί όπως θα ακούσετε, σήμερα ήδη κάνει επιλογή εκστρατεία. Έχει δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, το κόμμα για τον Brexit, για να προσπαθήσει να υπερκεράσει τους συντηρητικούς. Και τα δύο μεγάλα κόμματα, η συντηρητική και η εργατική, υπάρχει κίνδυνος να υποστούν τεράστια ήττα στις ε, ευρωεκλογές. Η συμβουλή μου λοιπόν προ αυτά τα δύο κόμματα είναι αν δεν είναι ανόητα κόμματα πρέπει να καταλήξουν συμφωνία τι επόμενε μέρε για να αποφευθεί αυτή η καταστροφή. Και κύριε Τάσκ, την επαύριο αυτή τη απόφαση είπατε κάτι το οποίο επαναλάβατε και τώρα πριν από λίγο. Είπατε ότι μπορεί να αποφύγουμε την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και κοιτάξτε, και εγώ είμαι κατά τη αποχώρηση, αλλά δεν είναι δική μα απόφαση. Είναι απόφαση του Βρετανικού λαού. Φόβο μου λοιπόν είναι ότι αντί να σκοτώσουμε τον Brexit, η απόφαση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο θανάτου για την Ευρώπη. Δηλαδή να βαλτώσουμε και πάλι για χρόνια. Όλη η ενέργειά μα να πηγαίνει σε διαπραγματεύσει με του Βρετανού ηγέτε. Όπω ο κύριο Κόρμπιν ή ο κύριο Τζόνσον. Οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι κατά τη Ευρώπη. Τη συχαίνονται. Ενώ χρειαζόμαστε όλοι μα την ενέργεια για να μεταρρυθμίσουμε, για να ανεώσουμε την ε, ε, δική μα Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό Πρέπει και εσείς να εστιάσετε ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε αυτά. Και αυτού του είδους η προσέγγιση ήταν απούσα κατά τη γνώμη μου την περασμένη Τετάρτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Τσίμερ, παρακαλώ δύο λεπτά. Κυρίες και κύριοι, Υπάρχουν στιγμές νομίζω που οι αντιπαραθέσεις ε, για τις εκλογές πρέπει να σταματούν. Μας έδειξε, έχετε χτεσινή για στο Παρίσι, πόσο ευάλωτος είναι ο κόσμος μας, πόσο εύθραυστη η Ευρώπη, ο πολιτισμός, η ιστορία και το μέλλον μας μαζί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη. Η Παναγία των Παρισίων είναι σύμβολο, σύμβολο της Ευρώπης, σύμβολο της Γαλλίας. Εγώ πριν από πολλά χρόνια Ανατολικό Ανατολικογερμανίδα ξεκίνησα να μαθαίνω γαλλικά και ήξερα ότι θα μπορώ να έρθω να δω την Παναγία των Παρισίων. Είναι μεγάλο το σοκ λοιπόν για όλους μας εδώ, τους συναδέλφους. Και λέμε σε όλους τους Γάλλους ότι είμαστε στο πλευρό σας, αλλά ταυτόχρονα απαιτούμε να αναγνωριστεί πόσο ευαίσθητο, ευάλωτο είναι όλο αυτό αυτή η πολιτιστική κληρονομιά όπως και η Ευρώπη και με πόση προσοχή πρέπει να την αντιμετώπισουμε. Ούτε εγώ είμαι ικανοποιημένη από την έκβαση και τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής. Βρίσκω ότι είναι μοιραία απόφαση αυτή που ελήφθη. Γιατί ό,τι απόφαση να έκβαση και, σημαίνει και αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται δεσμευμένο σε μια τέτοια ε, εξέλιξη επί ένα εξάμεινο. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα γίνουν οι εκλογές, θα περάσει η θερινή περίοδος, θα αρχίσουν οι ε, συγκροτήσεις ομάδων και κοινοβουλίου, θα είναι οι Βρετανοί μέσα ή έξω, θα έχουμε να ε, σχέδιο Α, ένα σχέδιο Β, θα λέμε ότι έχουμε επιτροπές με μέλη τάδε και τάδε, πρόεδρου τάδε και δίνα, αλλά στην περίπτωση που θα υπάρχουν οι άλλοι, θα ε, υπάρχει διαφορετική σύνθεση ή και δύναμη των ομάδων. Έχετε σκεφτεί τι είναι αυτό με το οποίο μπορούμε να συνερπάσουμε τον πολίτη για την Ευρώπη σήμερα. Ήδη είναι τόσο δύσκολο όταν ξέρουμε ότι εκ των προτέρων βλέπει ένα τσίρκο ο πολίτης. Είναι δυνατόν να, μην, να δεσμεύεται το κοινοβούλιο για, την επόμενη, για τους επόμενους μήνες και να μην είναι ξεκάθαρη κατάσταση για όλη τη θητεία. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κυρία Σκοτκάτο, ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, έφτασε Πάσχα και είμαστε ακόμα εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερος και εγώ και τα εκατομμύρια των Βρετανών συμπολιτών μου. Χαίρομαι που μπορώ να ολοκληρώσω τη θητεία που μου εμπιστεύτηκαν οι ψηφοφόροι της Νοτιοανατολικής Αγγλίας και του Γιβραλτάρ πριν από πέντε χρόνια. Εμείς αυτό το εξάμεινο θα το αξιοποιήσουμε. Εμείς οι πράσινοι την προκλογική εκστρατεία θα την αξιοποιήσουμε για να προβάλλουμε τις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είμαστε μια από τις πιο ισχυρές δυνάμεις και θα υπερασπιστούμε στην Ευρώπη μια, μια πιο πράσινη Ευρώπη, μια πιο δημοκρατική και πιο ισχυρή Ευρώπη και ευχαριστώ τον πρόεδρο Τούσκ που μας έδωσε αυτό το περιθώριο να πάρουμε μια ανάσα και να ξανασχεδιάσουμε το μέλλον μας. Ποτέ δεν ήταν ευχερή η οικοδόμηση της Ευρώπης. Ο κύριος Τούσκ παρέπεμψε στο ιστορικό και τους ιδρυτές της Ευρώπης οι οποίοι έκαναν προσπάθειες για να συμπεριλάβουν και να κρατήσουν μέσα στην Ευρώπη αυτού που είχαν και στο εσωτερικό τους, στο εσωτερικό της χώρας τους εγώ ως πράσινη πάντοτε ήμουν σκληρή η επικρίτρια του Brexit, αλλά πρέπει να είμαστε σκληροί επικριτές και στα αίτια που οδήγησαν στο Brexit. Δηλαδή την ιδέα που έχει ο πολίτης ότι είναι αδύναμος, ότι έχει απομακρυνθεί, ότι δεν έχει κανένα λόγο στην Ευρώπη. Και αυτό οδήγησε στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2016. Για εκείνους λοιπόν τους φίλους οι οποίοι ήταν υπέρ της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου, το μήνυμα ήταν, είναι ας αξιοποιήσουμε αυτό που υπάρχει, ας προβάλλουμε τα καλά της Ευρώπης, ας καταρρύψουμε τις ειρήνες των ακροδεξιών. Πρέπει με τις επόμενες εκλογές να κερδίσουμε την ψήφο του πολίτη, να πείσουμε τον πολίτη, τον συμπολίτη μας ότι το καλύτερο μέλλον για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι να παραμείνει κομμάτι αυτής της ευρωπαϊκής οικογένειας. Mr. Farage, five minutes. Thank you. Good morning. Well, I have tried for 20 years Κοιτάξτε, εδώ και 20 χρόνια προσπαθώ να φύγω από εδώ πέρα. Και νόμιζα ότι είχα πετύχει. Αλλά δεν είχα καταλάβει τι θα έκανε η πολιτική τάξη του Ηνωμένου Βασιλείου. Και κοιτάξτε, το μήνυμά μου είναι θα ξανάρθω. Πολλοί από εμά θα ξανάρθουν. Γιατί ο κύριο Φερχόφστατ έχει δίκιο. Ναι, ναι, το είπα. Ναι, ήμουν ο πρώτο που το είπα αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το κόμμα του Brexit θα σκίσει σε αυτέ τι εκλογέ. Και μόνο ένα τρόπο είναι να το σταματήσετε. Είναι το κόμμα τη κυρία Μέη και η αντιπολίτευση του κυρίου Κόρμπιν να συμφωνήσουν και να συμφωνήσουν σε μια μόνιμη τελεωνική ένωση και στην ουσία ε, να είναι και μέλη τη ενίας αγορά. Αν γίνει αυτό, το κόμμα του Brexit δεν θα κερδίσει τι ευρωεκλογέ. Θα κερδίσει τι εθνικέ εκλογέ. Γιατί η προδοσία θα είναι τόσο ολοκληρωμένη και καταφανή. Δεν νομίζω γι' αυτό ότι θα συμβεί αυτό. 15 χρόνια που είμαι πρόεδρος ε, ε, με άλλους ή μόνος μου ενός πολιτικού κόμματος, έχω συμμετέχει, συμμετάσχει σε πολλές συναντήσεις κορυφής και έχω δει πολλές συγκρούσεις μεταξύ κρατών και των ευρωπαϊκών ε, θεσμών, η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία ή η Ελλάδα. Και υπάρχει ένας χρυσός κανόνας. Πάντα. Είναι ότι κερδίζει οι Βρυξέλλες. Η ισχύ των Βρυξελών τα καταφέρνει πάντα να κερδίσει. Αλλά ποτέ δεν πήγα σε συνάντηση κορυφή όπως την προηγούμενη εβδομάδα όπου για δεύτερη φορά σε δύο εβδομάδες μια Βρετανίδα πρωθυπουργό έρχεται και ζητιανεύει, ζητιανεύει. Παρακαλά για μια παράταση του άρθρου 50. Ήταν ξεφτύλα. Όχι μόνο να είναι κανεί στι Βρυξέλλε. Ξεφτύλα, ταπεινωτικό για τη χώρα μα. Την θέση τη στον κόσμο. Ξέρετε, έχουμε την κοινοπολιτεία, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχουν πολλέ χώρε που μα γουστάρουν. Θεωρούν ότι είμαστε ακόμα ένα μεγάλο έθνο. Και όμω έχουμε πέσει τόσο χαμηλά. Η Πρωθυπουργό που μα υποσχέθηκε ότι θα φύγουμε στι 29 Μαρτίου είπε ε, μπορεί να φύγουμε στις 12 Απριλίου. Θα φύγουμε οπωσδήποτε στις 30 Ιουνίου. Και τώρα τι μας λέει. Θα φύγουμε 31 Οκτωβρίου. Θα είναι Halloween δηλαδή. Ή γλυκό ή φάρσα. Ε, ελπίζω, ελπίζω να αποχωρήσουμε τελικά. Αλλά αν το αφήσουμε σε αυτή την άθλια πρωθυπουργό αν αφήσουμε του ε, πολιτικού μα στο κοινοβούλιο να χειριστούν το θέμα, δεν θα συμβεί ούτε αυτό. Στο παρελθόν ξέρω ότι πάντα επέκρινα τη δύναμη χωρί λογοδοσία των ε, κυρίων ε, γραφειοκρατών των Βρυξελών. Αλλά πρέπει αυτή τη φορά να πω ότι για αυτά τα χάλια δεν φταίτε εσεί. Από την αρχή είχατε σαφή θέση. Αυτά τα χάλια είναι ευθύνη των δύο μεγάλων βρετανικών κομμάτων που και τα δύο μας υποσχέθηκαν στα προεκλογικά τους προγράμματα ότι θα υπάρξει Brexit που δέχθηκαν να πυροδοτηθεί το άρθρο 50 που είπαν ότι θα φύγουμε με συμφωνία χωρίς. Μας πρόδωσαν, αυτοί μας πρόδωσαν. Και συμφωνώ την, ε, με τη θλίψη που εξέφρασαν και οι άλλοι για την καταστροφή χθε της Νόρνταν. Κάτι τόσο όμορφο καταστράφηκε αλλά ε, χάνεται και κάτι άλλο πολύ ζωτικό για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και νομίζω ότι χθε ε, οι νεκρολογίε του Times το έλεγαν. Πολύ σωστά. Ε, η νεκρολογία έλεγε ότι η δημοκρατία του Ηνωμένου Βασιλείου 312 ετών πέθανε στις 29 Μαΐου. Πέθανε ίσχα στον ύπνο της στις 11 το απόγευμα στις 29 Μαρτίου 2019. Αιτία θανάτου, δολοφονία και οι ένοχοι ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί. Η δημοκρατία ε, ήταν ε, κάτι το οποίο στήριζε ε, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αποφάσεις. Θα μας λείψει ο Θεός να μας βοηθήσει. Αυτό που θα γίνει στις 23 Μαΐου δεν έχει να κάνει μόνο με τον Brexit και την αποχώρησή μας από την Ένωση. Είναι για το τι είδους χώρα είμαστε. Έχουμε την παλιότερη κοινοβουλευτική παράδοση στον κόσμο. Τη μητέρα των κοινοβουλίων. Αγωνιστήκαμε και δώσαμε πολλά για αυτή την αρχή τη δημοκρατία ενό εθνικού κράτου, όχι μόνο για εμά, αλλά για του φίλου μα στην Ευρώπη. Και ορισμένοι εδώ, στη χώρα μου μάλλον καλύτερα, είναι απογοητευμένοι. Αλλά άλλοι είναι τρομερά αγανακτισμένοι. Δεν βάζουν κίτρινα γυλαίκα εκείνοι. Αλλά λένε, χρειαζόμαστε μια ειρηνική πολιτική επανάσταση στη χώρα μου. Πρέπει να εξαφανιστούν τα δύο αυτά κόμματα τα οποία μας πρόδωσαν. Και νομίζω ότι όλοι σας θα εκπλαγείτε ιδιαίτερα από αυτά που θα συμβούν στις 23 Μαΐου. Θα είναι μια καινούργια αρχή για τη Βρετανική Δημοκρατία και πραγματικά τη χρειαζόμαστε. Συνάδελφοι, λέει πρόεδρος, έλαβα κάποια αιτήματα για μπλε κάρτα, αλλά επειδή Υπάρχει ήδη προηγούμενο, δεν υπάρχουν μπλε κάρτε κατά τη διάρκεια τη συζήτηση των ηγετών. Και τώρα ο κύριο Μπάτεν, τρία λεπτά. Όλα αυτά δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβαίνουν αν είχε τιμηθεί η απόφαση του δημοψηφίσματος το 2016 και η Βρετανία είχε φύγει εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, η δημοκρατική απόφαση 17,4 εκατομμυρίων ανθρώπων η θελημένα προδίδεται. Οι ευρωεκλογέ του Μαΐου αναπόφευκτα θα είναι μια επανάληψη του δημοψηφίσματος. Όποιο, ό,τι και αν πούνε τα πολιτικά κόμματα, η επιλογή των ψηφοφόρων θα είναι στην ουσία επί του αν θα μείνουμε ή θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ του να μείνουμε θα πρέπει να ψηφίσουν τους ε, φιλελεύθερους δημοκράτες. Είναι το κόμμα του παραμένουμε. Ενώ αυτοί που θέλουν να φύγουν θα πρέπει να, ψηφίσουν το κόμμα της ε, ανεξαρτησίας. Το UKIP είναι ε, το κόμμα που θα προχωρήσει στην έξοδο. Οι υπόλοιποι δεν ξέρουν ούτε καν τι θέση έχουν για αυτό το θέμα. Η πολιτική του UKIP είναι σαφής ε, και ξεκάθαρη. Είναι της μονομερούς και ανεφόρων εξόδου. Αυτές όμως οι εκλογές θα διχάσουν τον κόσμο σε δύο διακριτές ομάδες, όχι μόνο σε Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η μια ομάδα θα είναι αυτή που συγκατατίθεται να τους κυβερνεί να μια ξένη δύναμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη ομάδα θα είναι αυτή που επιλέγουν να επαναστατήσουν ενάντια σε περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και υπέρ της επιστροφής των δημοκρατικών ε, αξουσιών στα κράτη-έθνη. Η μια ομάδα θα αγωνίζεται για την ελευθερία και την ανεξαρτησία, η άλλη ομάδα θα ψηφίσει υπέρ της υποδούλωσης και της υποταγής. Κάτι για το οποίο ε, ε, πρέπει να είμαστε βέβαιοι είναι ότι οι ευρωσκεπτικιστέ, οι ευρωβουλευτέ θα επανέλθουν πολύ ε, άριθμοι, πολύ άριθμοι και οι ψηφοφόροι τους θα ψηφίσουν υπέρ της επιστροφής στη δημοκρατική λογοδοσία στο τέλος των μέτρων λιτότητας και στην διαχείριση των οικονομιών προς το συμφέρον τους και το όφελό τους θα ψηφίσουν υπέρ τη πάυση τη μαζική και ανεξέλεγκτη μετανάστευση. Θα ψηφίσουν υπέρ κομμάτων που θέλουν να διατηρήσουν τον πολιτισμό του και την κουλτούρα του. Και θα το, το UKIP θα, είναι η ψήφο, η λαϊκή ψήφο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε την ψήφο υπέρ του παραμένουμε ή του υπέρ του φεύγουμε οι ε, εκλογέ τις οποίες παρότρινε το UKIP έφεραν το δημοψήφισμα και το UKIP θα εξακολουθήσει τον αγώνα ώστε να γίνει πραγματικότητα το Brexit. Στις 31 Μαΐου οι βουλευτές που θα, του UKIP θα συνεχίσουν τον πολιτικό αγώνα ώστε να απελευθερωθεί το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία ψήφος υπέρ του UKIP στις 31 Μαΐου θα στείλει σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση να φύγουμε και από το ΠΟΕ άμεσα. Το UKIP δεν είναι μόνο μια εκστρατεία υπέρ του Brexit. Θέλουμε αυτό να γίνει πραγματικότητα. Μια ψήφο στο UKIP σημαίνει πάντα αποχώρηση από την, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι Βρετανοί θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ του UKIP στις 31 Μαΐου. Ο κύριος και ένα λεπτό παρακαλώ. Μια εγγεγραμμένος. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισιών στις Φλόγες ήταν ε, εικόνα τραγική. Όλοι βέβαια, υπόθηκε νωρίτερα, πρέπει να αντιληφθούμε ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να λάβουμε τις δύσκολες αποφάσεις. Καλωσορίζω την απόφαση του Συμβουλίου για την παράταση της προθεσμίας του Brexit. Απεφεύχθη το μοιραίο, η σύγκρουση. Μόνο αυτοί που, μόνο αυτοί που είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και του Ηνωμένου Βασιλείου ε, είναι δυσαρεστημένοι. Και βέβαια ο κύριος Φαράζ δεν με ξάφνιασε. Με ξάφνιασε όμως ο κύριος Φερχόφστατ, που φαίνεται φεντεραλιστής όν, να κάνει τη δουλειά των λαϊκιστών. Δηλαδή να λέει ότι πρέπει να φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο. Όχι, δεν είναι αυτή η λύση. Χρειάζεται πραγματισμό, ρεαλισμό, συνεργασία. Ελπίζω με την προσεχή ε, περίοδο τη βουλευτική να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτό. κύριο Μπροκ, ένα λεπτό και 30 δεύτερα. Πρόεδρε, Πρόεδρε του Συμβουλίου, Πρόεδρε τη Επιτροπή, αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχουμε νέα κατάσταση, νέε συνθήκε τον Οκτώβριο ή θα ξαναζούμε την ίδια κατάσταση με αυτή που έχουμε σήμερα γιατί θα έχει το ζήτημα. Ελπίζω να βρούνε μια λύση ο Κόρμπιν και η Μέη. Να πιέσουν το, τη Βουλή των Κοινοτήτων να βρούνε μια επικοδομητική λύση είτε για να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε για να αποχωρήσουν πάντως όχι με ε, μεσοβέζικες λύσεις, λύσεις και πρέπει εμείς να κοιτάξουμε πλέον να ασχοληθούμε με τα μεγάλα προβλήματα που μας περιμένουν στο μέλλον, τα ζητήματα της μετανάστευσης, των πολέμων των εμπορικών συναλλαγών, των, ε, της ασφάλειας, τα εξωτερικά σύνορα, σύνορα της κλιματικής αλλαγής και πολλά άλλα. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη δύναμη με την οποία μπορούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τις, μεγά, τις μεγάλες απειλές των Τραμπ και των του, Πούτιν του κόσμου και να σώσουμε έτσι την Ευρώπη και να τις επιτρέψουμε επιτρέψουμε να προοδεύσει. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε ως μια μεγάλη δύναμη και να μην επιτρέψουμε το διχασμό που φέρνει ο λαϊκισμός. Έτσι λοιπόν με την Ευρώπη αυτή, την Ευρώπη της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της ελευθερίας, της ανθρωπιάς, της ε, επιτυχίας της Ευρώπης αυτής ε, η οποία έχει εξασφαλίσει τόσα πολλά για όλο τον κόσμο, για όλους τους πολίτες. Ύστερα από 39 χρόνια η τελευταία μου ομιλία είναι η σημερινή και με αυτήν θέλω να σημειώσω ότι η Ευρώπη στέφθημε με επιτυχία στην ιστορία της ε, ανθρωπότητας. Σε νέα κράτη ήμασταν όταν εγώ πρωτοέγινα βουλευτής. Ε, και δεν λειτουργούσε ακόμα καλά-καλά η Τελωνιακή Ένωση. Τώρα έχουμε φτάσει στα 28 κράτη-μέλη και πρέπει αυτή την ένωση να την τιμήσουμε και να ε, εξηγήσουμε και στον πολίτη, στον ψηφοφόρο γιατί είναι τόσο σημαντική. Μπορεί να μην είναι μόνο ένα ωραίο ε, κτίριο ή ναός η Παναγία των Παρισίων είναι πολιτιστική κληρονομιά πάνω από όλα, όχι μόνο της Γαλλίας αλλά όλης της Ευρώπης και όλου του κόσμου και θυμάμαι τη στιγμή εκείνη που Κάναμε την επιμνημόσυνο δέηση για τον Helmut Kohl, ε, με τον Helmut Kohl για τον François Mitterrand. Είναι η στιγμή η οποία δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς, μια στιγμή ενότητας και ήρθε ο Φρανσουά Μιτερό εδώ στο Κοινοβούλιο για να πει λέει συγκινημένο ο ομιλητή, ότι ο, ο εθνικισμό ε, ισοδυναμεί με πόλεμο. Αυτά τα λόγια δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε ποτέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπροκ. Είναι τελευταία σας ομιλία στο σώμα μας. Υπηρετήσατε ιδιαίτερα καλά το σώμα και ελπίζω να μην ξεχάσετε τελώ την ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα θα την αντιμετωπίζετε από άλλη οπτική γωνία. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι το σώμα απέτυσε φοροτιμής με το χειροκρότημά του σε εσά. It's one of those emotional ε, κύριε Μπρόκ, ε, υπάρχει πολύ συγκινησιακή φόρτιση ε, σήμερα το πρωί και νομίζω ότι διαπιστώνετε σε εκτιμούν οι συνάδελφοί σα. Ο κύριο Κόρμπετ, τώρα για δύο λεπτά, ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με όσου αναφέρθηκαν στην τραγωδία του Νότρο Ντάμ και ιδιαίτερα αυτά που είπατε εσεί ότι και εμείς συμμεριζόμεθα τον πόνο του γαλλικού λαού. Είπατε ότι δεν μα συνδέουν απλώς συνθήκες και κείμενα. Αυτό ισχύει. Και γι' αυτό ε, σκανδαλίστηκα όταν τη στιγμή που το λέγατε αυτό ο κύριος Φαράτζ, ο οποίος έχει ήδη φύγει ως συνήθως, φώναξε βλακίες. Αυτό νομίζω ότι αποδεικνύει τη στάση πολλών από την άλλη πλευρά. Αλλά είναι η φωνή του παρελθόντος. Ο Βρετανικός λόγος αρχίζει να καταλαβαίνει τι ψέματα του λένε εδώ και χρόνια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίζουν να βλέπουν τα ψέματα που του είπατε για τον Brexit. Μα είπατε ότι θα ήταν πολύ εύκολο. Ε, είναι αρκετά περίπλοκο, ε. Μα είπατε ότι θα εξοικονομούσαμε πολλά χρήματα για το σύστημα υγεία μα. Τελικά θα μα κοστίσει μια περιουσία. Μα είπατε ότι θα έχουμε έτοιμε νέε εμπορικέ συμφωνίε με χώρε παντού στον κόσμο για να αντικαταστήσουν ε, το εμπόριο που θα χάσουμε από την Ευρώπη. Χάνουμε όλε τι ε, συμφωνίε που έχουμε μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αν υπάρξει Brexit. Ο Βρετανικό λαό αρχίζει να αντιλαμβάνεται τι του είπαν. Και γι' αυτό φοβούνται τόσο πολύ το να γίνει ένα νέο δημοψήφισμα. Γιατί ξέρουν ποια θα ήταν η απάντηση αν υπήρχε νέο δημοψήφισμα. Γι' αυτό οι συντηρητικοί δεν θέλουν να γίνουν ευρωεκλογέ. Γιατί ξέρουν ότι θα συντριβούν σε αυτέ τι εκλογέ. Και εκπλήσω με λιγάκι που ο κύριο Φερχόφστατ και ορισμένοι άλλοι εδώ στο σώμα μα, εδώ φοβούνται αυτέ τι εκλογέ. Γιατί φοβάστε, δεν υπάρχει λόγο. Η πλειονότητα των ευρωβουλευτών που θα επιστρέψουν δεν θα είναι του φυράματος των απέναντι. Και, εν πάση περιπτώσει, εν πάση περιπτώσει, το Brexit, η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενός μέλους για πρώτη φορά, οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης είναι πολύ πιο σημαντικές από το συσχετισμό δυνάμεων των πολιτικών ομάδων Δείτε τα πράγματα στο σωστό πλαίσιο. Αυτή η παράταση πρέπει να αξιοποιηθεί όπως σωστά είπε ο κ. Τούσκ. Εντάξει, δεν έχω και πολλές ε, μεγάλες προσδοκίες για ε, τη συζήτηση μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων. Γιατί η κυρία Μέη δεν μπορεί να αλλάξει θέση χωρί να αντιμετωπίσει ανταρσία από το κόμμα τη, αλλά μα δίνει μια ευκαιρία να επανέλθουμε στο λαό και να σταματήσει αυτό το άθλιο χάλι στο οποίο έχουμε καταλήξει. Ευχαριστώ πολύ.